συναδέλφους οι οποίοι έχουν εργαστεί πολύ σοβαρά στην κατάρτιση αυτών των τροπολογιών. Το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές τροπολογίες εγώ θεωρώ ότι είναι ένα θετικό στοιχείο. Δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα για να υπάρχει μία ικανοποιητική πολιτική αλληλείας η οποία πρέπει να οργανωθεί σωστά Γι' αυτό και αναγνώρισα τους συντάκτες ορισμένων τροπολογιών και ελπίζω θα καταφέρουμε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα το οποίο περιμένω. Ευχαριστώ κύριε Ρόντας. Ευχαριστώ για όλη την εργασία την οποία έχετε κάνει επί του θέματος. Έχω διαβάσει εκατοντάδες από τις τροπολογίες κατά τις διακοπές και έχω πλήρη κατανόηση για αυτά που είπατε. Ελπίζω ότι οι σκιώδεις εισηγητές στις τέσσερις συνεδριάσεις που αναφέρατε θα μπορέσουν να συνοψίσουν τις τροπολογίες αυτές σε ε, τροπολογίες ε, οι οποίες θα γίνουν ε, κοινά αποδεκτές, διαφορετικά θα ψηφίζουμε ως τα Χριστούγεννα ε, η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ κατά το καλοκαίρι εξέτασα με λιγότερο ζήλο ίσως από την κυρία Ρόντου στο, την πληθώρα των τροπολογιών που υπευλήθησαν από τους συναδέλφους. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκες και ακολουθούν όλες τις δυνατές κατευθύνσεις αυτό που είναι σημασία δεν είναι τόσο πολύ οι τροπολογίες διότι και εμείς θα πρέπει να τις συζητήσουμε στα πλαίσια των πολιτικών ομάδων όπου επίσης διήστανται οι απόψεις αλλά πρέπει να οριοθετήσουμε τη συζήτηση διότι το βασικό είναι το αποτέλεσμα και πρέπει να επιτύχουμε ένα ως το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα για την κοινή αλληλευτική πολιτική στην κυρία Ρόντουστ η οποία λέγει ότι έχει στείλει ηλεκτρονικά μηνύματα πρέπει να πω ότι εγώ δεν έχω λάβει τίποτα άρα δεν μπορώ να σχολιάσω τις συμβιβαστικές τροπολογίες της κυρίας Ρόντουστ και επιπλέον για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις συμβιβαστικές πρέπει να έχουμε μια συνολική επισκόπηση, δηλαδή να έχουμε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να εργάζομαι με τρόπο κατακαιρματισμένο. Χρειάζομαι το σύνολο των συμβιβαστικών τροπολογιών και θα ήθελα να μπορέσουμε να αναλύσουμε γενικά όλες τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες που έχετε καταρτήσει διότι δεν θα υπογράψω μία επιταγή εν λευκό αν δεν έχω μία συνολική εικόνα. Αυτή είναι η πρόταση εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδος. Έχετε προτείνει τέσσερις ε, ε, συναντήσεις. Ο τομέας της αλληλείας περιμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αποτελέσματα αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η βία να, για να καταλήξουμε σε ένα ε, κακό αποτέλεσμα. Μακάρι να τα καταφέρουμε και να συμφωνήσουμε σε τέσσερις συνεδριάσεις. Όπως είπε η κυρία Ρόντους, μπορούμε να συνεργαστούμε και πέραν αυτού του χρονοδιαγράφωνος. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε επί του θέματος αυτού, αλλά το βασικό κατ' εμέ είναι πρώτα απ' όλα να έχουμε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Δεύτερον, να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και αν ε, δεν ικανοποιηθούμε θα χρειαστεί ίσως και περισσότερος χρόνος. Αυτό που είναι βασικό είναι να μπορέσουμε προς το παρόν να σχολιάσουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα εφόσον δεν έχω τα έγγραφα εργασίας. Η προσωπική μου θέση υπάρχει στις τροπολογίες μου, δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσω εδώ. Ξέρει η κυρία Ρόντους τι σκέφτομαι, αλλά θέλω να ξέρω αν για την περιφερειοποίηση έχουμε καταλήξει σε κάποια τροπολογία, γιατί αυτό θα είναι το πιο δύσκολο να ρυθμιστεί σωστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω, έχω καταλήξει. κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Ρόντου, τον συγγήτρια. Καταλαβαίνω ότι έκανε πολλή δουλειά μέσα στο καλοκαίρι. Δυσκολήθηκα και εγώ ώρες, για να μην πω ημέρες, με τις τροπολογίες και οφείλω να πω ότι συμφωνώ με τόσο είπε η κυρία ότι είναι τόσες πολλές οι ταυτόσιμες ε, τροπολογίες που θα ήταν σωστό να γίνει μια προσπάθεια να τις ε, ενοποιήσουμε, να τις ομαδοποιήσουμε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και μια και είναι πολλές οι τροπολογίες, που κοιτάξαμε σε πολλά ουσιαστικά σημεία τους ε, στις συζητήσεις επιτροπής. Δεν θεωρώ σκόπιμο να αρχίσει η συζήτηση για τα θέματα επί της ουσίας δηλαδή πριν να δούμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Είναι δύσκολο αυτό. Ξέρω ότι έχουμε πολλά θέματα να καλύψουμε. Πάντως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ομάδα μας, η ομάδα των Πρασίνων, είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί και να εργαστεί σκληρά μαζί με όλους τους κοιόδης, τους, ε, την συγκήτρια. Η κυρία Φράγκα βεβαίως εύστοχα επισημαίνει ότι καλό θα ήταν να δούμε όλες τις ε, συμβαστικές τροπολογίες για να έχουμε μια γενική εικόνα. Αλλά εμείς θα ακολουθήσουμε την εισηγήτρια σε όποια μέθοδο προτείνει. Έστω και αν δεν την έχουμε δει λεπτομερώς ακόμη. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χάτσιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια που μας περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα. Φιλόδοξο πρέπει να πω, δεδομένου και του όγκου της ύλη που έχουμε να επεξεργαστούμε. Πριν από 10 χρόνια περίπου που είχαμε αντίστοιχες συνεδριάσεις που είχαμε περάσει μέρες με συμβαστικές ε, συζητήσεις με τροπολογίες που είχαμε θεωρήσει τότε πάρα πολλές αλλά δεν συγκρίνονται σε τι, με, με, ε, είναι αυτές που έχουμε τώρα να διαπραγματευτούμε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να συνεργαστούμε στην συνεδρία των σκιωδών για τις συμβαστικές τροπολογίες. Γιατί ναι, μα πιέζει ο χρόνο και πρέπει να γίνει δουλειά, αλλά η κύρια ευθύνη μα, η σημαντικότερη ευθύνη μα είναι να γίνει σωστά η δουλειά αυτή τη φορά. Και για να επαναλάβουμε ενδεχομένω ε, την συζήτηση που είχε γίνει κατά την εισαγωγή του θέματος αυτού πριν από μερικά χρόνια αν υπενθυμίσω, και να υπενθυμίσω ότι είχε χαρακτηριστεί ως αποτυχία η προσέγγιση που είχε ακολουθηθεί θα ήθελα να πω ότι τώρα πρέπει να βρούμε τη σωστή λύση, έστω και αν χρειάζεται να τροποποιήσουμε ελαφρώ το χρονοδιάγραμμα ή να βρούμε εναλλακτικέ. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να ζητηθούν λόγοι για καθυστέρηση, αλλά υπάρχουν δυνατότητες, έχουμε μέσα στα χέρια μας και πρέπει χάρη σε αυτά να κάνουμε καλή δουλειά. Αν ε, ήταν να σχεδιάσουμε την πολιτική για τη διαχείριση των ελευτικών αποθεμάτων. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Θα, πρέπει να ξεκινήσουμε από μια τάμπουλα ράζα. Και γι' αυτό νομίζω ε, μια από τι πιο σημαντικέ τροπολογίε, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην συζήτηση αυτή θα πρέπει να είναι η αποκέντρωση, η ο εξυγχρονισμό, όπω αλλιώ το πούμε, Οτιδήποτε δηλαδή χρειάζεται ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και να επιτευχθεί πιο καλό επίπεδο λήψεως αποφάσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ενθουσιασμού θα τα χαρακτήριζα ως προς το μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Οι 100 τόσες δικές μου αποτελούν μόνο κλάσμα του συνόλου εγώ πάντως επιμένω στην αποκέντρωση, διότι θεωρώ ότι με το να αποκεντρώσουμε την ουσιαστική εξουσία στην ε, αλία και με το να δώσουμε πραγματική ε, εξουσία λήψης αποφάσεων σε εκείνους που κερδίζουν από τη ζωή τους από την αλία θα είναι ο καλύτερος τρόπος για καλές αποφάσεις, για σωστές λύσεις. Και γι' αυτό αντιδρώσω μέσα από τι αρχικέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίε επιβάλλουν ε, μια κεντρική διαχείριση σε μεγάλο βαθμό μέσα από το πλαίσιο που προτείνεται και όχι την αποκέντρωση. Γι' αυτό και προτείνω και στη διατύπωση ακόμη τροποποίηση το ΣΑΛ ή το ΜΕΙ, εκεί που γίνεται λόγος για τις δυνατότητες ε, εισαγωγή μέτρων από τα κράτη-μέλη, είναι ήδη μια συγκεκριμένη επιλογή και έχει σημειολογική βαρύτητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέρη να συνεργαστούν με τρόπο λογικό στις θαλάσσιες λεκάνες εκείνες όπου ο εμπλεκόμενος ή εμπλεκόμενοι αλληλείς, οι παράγοντες της αλληλείας θα μπορούν να συνδιαμορφώσουν τις επιλογές για να διαφυλάξουν τα αλληλευτικά αποθέματα και τον βιοπορισμό των αλληλευτικών κοινοτήτων. Περιμένω λοιπόν να δω τι είδους συνεδριάσεις θα οργανώσουμε μαζί, θα συνοργανώσουμε και βεβαίως ελπίζω σε πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά για άλλη μια φορά απευθύνω έκκληση αυτή τη φορά να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει αποτελέσματα επιτυχή και όχι απλώς να επιδιώκουμε πηχαίους τίτλους εφημερίδες και ε, μια καταδικασμένη σε αποτυχία μέσα σε ορατό χρονικό διάστημα 5-10 χρόνια ε, λύση. Για να μην χρειαστεί μέσα σε 5-10 χρόνια να ξανασυζητήσουμε μια κοινή αλλιευτική πολιτική η οποία πάλι θα έχει ε, καταδικαστεί ως αποτυχημένη. Ευχαριστώ πολύ και ο τελευταίος εκ μέρους των σκιωδών είναι ο κύριος Φερέιρα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θεωρώ ότι τούτη τη στιγμή δεν μπορώ να προσθέσω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι χρήσιμο θα ήταν να έχουμε τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις επί της εκθέσεως αυτής. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω το εξής. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι πολύ συχνά σε σημαντικούς τομείς για τους οποίους ε, συζητούμε και σχετικά με τη μεταρρύθμιση της, πολιτικής της ε, πολιτικής, η θέση της Κομισιόν είναι αυτή η οποία τελικά ε, μπορεί να δώσει τον τόνο. Πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να εκριζώσει εντελώς της, ε, την κεντρική γραμμή των προτάσεων εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όμως εδώ ριζικά να αλλάξει η πρόταση. Η πρόταση της Κομισιόν βρίσκεται έτη φωτός μακριά από τις ανάγκες του τομέα ε, αλλά βεβαίως ε, εκείνη θέλει να συνεχίσει με την επικεντρωμένη πολιτική η οποία έδωσε τα τελευταία χρόνια ε, τα αποτελέσματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε δει τις τροπολογίες ε, και πιστεύουμε ότι η δυνατότητα να αντιταχθούμε ε, σε αυτήν την πρόταση τελικά είναι μειωμένη. Δεν έχουμε δυνατότητα να τροποποιήσουμε πλήρως την πρόταση αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάθε διάθεση, έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά με μεγάλο σκεπτικισμό αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο σοβαρών αποτελεσμάτων. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Είναι απαραίτητο το χρονοδιάγραμμα να ε, γίνει σεβαστό. γιατί παρότι υπάρχει επίγον χαρακτήρας θα πρέπει να σεβαστούμε τις ε, διάφορες, ε, τα διάφορα στάδια. Ο διάλογος, ε, η πορεία μας θα πρέπει να είναι καλά διαρθρωμένη και βεβαίως συμφωνώ και με αυτά που είπε και η συνάδελφος Φράγα. Η δημοκρατία έτσι είναι και απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. χρειάζεται, απαιτεί προσπάθεια και δουλειά το δημοκρατικό αποτέλεσμα. Ενδεχομένως κάποια πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει πιο πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, πρέπει να δουλέψουμε με συγκεκριμένο ε, χρονοδιάγραμμα. Και πάντως ε, να επαναλάβω αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι τα περιθώρια λιγμών του Κοινοβουλίου είναι μικρά. όσον αφορά τώρα τα την ε, δυνατότητα ας πούμε, που έχουμε όσον αφορά τα, τα μεταφερόμενα δικαιώματα, ε, ε βλέπουμε ότι είναι αρκετά πιεστική η πρόταση της ε, Επιτροπής. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε προηγουμένως ο συνάδελφος Χάτσον, ο γιατί πρέπει να έχουμε αποκέντρωση, αποκέντρωση και ξανά αποκέντρωση. Ε, τα αποτελέσματα, τα καλά αποτελέσματα της αποκεντρωμένης πολιτικής ε, τα έχουμε δει ήδη και πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να επαναλάβουμε αυτά που έγιναν τα τελευταία 30 ε, χρόνια και τα οποία βλέπουμε να επαναλαμβάνονται στην πρόταση της ε, Επιτροπής. Δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο ελιγμών παρά τις 2.500 τροπολογίες. Ε, θα συμφωνήσω με κάποιες από τις εκφράσεις σκεπτικισμού που έχουν αναφερθεί. Αλλά παρόλα αυτά βεβαίω με μεγάλη διάθεση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριο Ντέιβις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, φανταζόμουν από την αρχή ότι θα είναι μεγάλη συζήτηση και μακροσκελής ε, και βλέποντας όλα αυτά τα, χαρτιά τα καθοδήγησης που παίρνουμε στα ε, στα γραφεία μας ε, φοβούμε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει και η συγκήτρια λίγο να μας βοηθήσει. Εν πάση περιπτώσει, οι συμβιβασμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί και θα πρέπει να βασίζονται ε, στην ε, ε, απάντηση στις προσδοκίες των εμπλεκομένων φορέων. Θέλουμε την αλληλευτική πολιτική βεβαίως να είναι μακρόπνοη. Θέλουμε ανανέωση, να επιτρέπει την ανανέωση των ελευτικών αποθεμάτων και θέλουμε να δώσει νέα πνοή στην ε, αλλιευτική βιομηχανία. Αυτό δεν σημαίνει επομένως ότι θα πρέπει να εξευρεθούν οι ελάχιστοι κοινοί παρονομοστές, αλλά ε, συμφωνίες οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τα αιτήματα των εμπλεκομένων φορέων και αυτό που αναμένουμε όλοι σαν έκβαση από αυτήν την ε, συζήτηση. Και τελικά με λίγα λόγια μπορεί κανείς να εκφράσει τα πάντα. Ε, αφορά η μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής τελικά την επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών τη της μεγαλύτερης δυνατής αηφόρου ανάπτυξης. Βεβαίως θέλουμε να παραμείνουν τα γέλτζα αλλά το θέμα είναι ε, θέλουμε ε, να γίνει μέχρι το 2015. Επίσης, δεύτερη ερώτηση, Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα μειωθούν τα αλληλευτικά από θέματα ε, ε, διατηρώντας τα ε, βέβαια διατηρώντας τα πάνω, above, όπως λέει η πρόταση από τα μέγιστα ανανεώσιμα αλλιεύματα ή θέλουμε να δεχτούμε και λίγο πιο κάτω, γιατί διαφορετικά θα έχουμε δυσκολία να επιτύχουμε τους στόχους. τρίτων. Ξέρουμε ότι ε, το Συμβούλιο είναι λίγο διστακτικό γιατί λέει ναι θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους where possible ε, οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Ε, αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί θέλουν να βρουν ε, οδούς διαφυγής από νομικά δεσμευτικές αποφάσεις. Επίσης η, ε, ε, επίσης, ε, για να μπορέσουμε να βρούμε την, το, μέγιστο ανανεώσιμο αλίευμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ο πιο εύκολος τρόπος βεβαίως είναι να το επιτύχουμε κόβοντας, περικόπτοντας κατά πάρα πολύ τις 100 την αλιευτική δραστηριότητα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις γιατί αυτό το where possible μας αφήνει ε, πολύ σκεπτικούς. Και φαντάζομαι ότι ε, τον Δεκέμβριο θα βρουν, ε, ο κάθε υπουργό θα βρει τον τρόπο να χρησιμοποιήσει το where possible ε, για να δημιουργήσει έτσι κάποιες προϋποθέσεις που θα είναι καλές για τη χώρα του. Και μετά ο επόμενος Υπουργό θα, θα πει «Α, υπάρχει δεσμευτικό προηγούμενο, δεν μπορώ να κάνω κάτι». Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσει οι οποίες θα εισαχθούν εδώ θα είναι νομικά δεσμευτικές για τους ε, ε, υπουργούς. Έτσι το MSY να, είναι, ε, να επιτευχθεί σωστά. Και παραμένει και ένα άλλο ε, ε, ζήτημα. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν διασταυρούμενες ε, συμβιβαστικές λύσεις και στο Κοινοβούλιο. Και μην ξεχνούμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει κάποια στιγμή να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο. Εάν θέλει το Κοινοβούλιο να έχει κάποιες δυνατότητες επιτυχίας απέναντι στο Συμβούλιο θα πρέπει να μπει με δυνατά διαπραγματευτικά χαρτιά, με μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Όσον αφορά το where possible, ε, μήπως μπορούμε να ζητήσουμε ας πούμε από το Συμβούλιο να αντιστραφεί ε, το άχθος της απόδειξης, ε, δηλαδή να πούμε κάτι ως πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται except where impossible, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι απολύτως αδύνατο. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias. Yo quiero θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, για αυτήν την ε, μεγάλη προσπάθεια. Διάβασε σχεδόν 2.600 τροπολογίες, τις διάβασε, τις ανέλησε, τις συνέπτυξε έτσι ώστε να φτάσει σε συμβιβασμούς. Αυτό είναι πολύ καλή δουλειά. Ε, αλλά δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, γιατί καμιά φορά το τέλειο είναι εχθρός του καλού. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάποια ε, συμφωνία, ε, γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε τώρα την εισηγήτρια να έχει έτοιμη τη δέσμη των συμβιβαστικών ε, λύσεων. Θα πρέπει να της δώσουμε λίγο χρόνο, να έχουμε μια ευελιξία. Αυτό που είναι σημαντικό πάντως είναι η γενική προσανατολισμή. Η μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής θα πρέπει ε, να είναι πρώτα απ' όλα κοινή πολιτική. Εγώ συμφωνώ με την αποκέντρωση, αλλά αποκέντρωση δεν σημαίνει ή δεν πρέπει να σημάνει, να σημάνει επανεθνικοποίηση της αλληλευτικής πολιτικής. Μιλάμε για κοινή αλληλευτική πολιτική ε, και ο καθένας θα πρέπει να ε, κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Θέλουμε ε, να καλυφθεί κοινωνικά και οικονομικά ο τομέας από την κοινή αλληλευτική πολιτική. Τώρα, ε, το, η μέγιστη βιώσιμη αποδοτικότητα. Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να το επιτύχουμε και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εάν καθορίσουμε στόχο όμως, ε, θα πρέπει να έχουμε και έναν οδικό χάρτη και να έχουμε και τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ε, δεν θέλουμε απλώς να ζητήσουμε να δείξουν όλοι καλή θέληση για να το ε, επιτύχουν. Εάν έχουμε τα μέσα θα μπορέσουμε να ε, καθορίσουμε και τις ημερομηνίε, αλλά πρέπει να έχουμε τα μέσα γιατί εάν τα μέσα δεν είναι διαθέσιμα τότε ο νομοθέτης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός γιατί τελικά δεν μπορεί να κατηγορήσει για αποτυχία τον κλάδο εάν ο ίδιος δεν δίνει τα μέσα στον κλάδο για να επιτύχει η μεταρρύθμιση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι, σε τι θα βασίσουμε την μεταρρύθμιση. Ε, κάτι άλλο σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχει η εσωτερική αγορά που είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και η κοινή αλληλευτική πολιτική ε, δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση στους κανόνες της ε, εσωτερικής αγοράς. Δεν μπορεί να ξεχωριστεί, δεν μπορεί να είναι μόνος του ο τομέας της αλληλευτικής πολιτικής. Επομένως και το θέμα των προγραμμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, επίσης, ε, τα, ε, τα θέματα των παραλιευμάτων. Θα πρέπει να μειωθούν τα παραλιεύματα όσο γίνεται πιο πολύ, έτσι ώστε να μην έχουμε απορρίψεις θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μετρήσουμε άλλωστε το φαινόμενο αυτό των απορρίψεων. Ε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε παράλληλη ή ε, ε, παράνομη αγορά, αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε το θέμα των απορρίψεων των παραλιευμάτων. Επίσης, ε, το θέμα της αλληλείας μικρής κλίμακος, ε, ε, της ηχθειοκαλλιέργειας μικρής κλίμακος επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά πολλές παράκτιες περιοχές και θίγει την τοπική οικονομία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ουσιαστικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο βεβαίως και για το περιβάλλον και για το τοπίο και νομίζω ότι στην ε, μεταρρύθμιση της κοινής ελευτικής πολιτικής θα πρέπει ένα κεφάλαιο να αφιερωθεί σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θέλω να ε, σχολιάσω. Καταρχήν, όταν το Συμβούλιο τον Ιούνιο ε, αποφάσισε ε, ότι θα μπορούσε να ε, υπάρξει ε, ένα θέμα με την βιομάζα μέχρι το 2020 δεν είχα αντιληφθεί ότι μιλούσαν για κάτι διαφορετικό. Εμείς εννοούσαμε το FMS μέχρι το 2015 και δεν είναι αυτός ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι όμως κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε κατά την συζήτηση των τροπολογιών και πρέπει εδώ να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις, διότι πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό και τι δεν είναι εφικτό διότι εάν ε, υπάρχει ε, μια βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων μέχρι το 2020 εκτός ε, από τον Βακαλάο τότε ενδέχεται να μην έχουμε επιτύχει με και ε, το στόχο μας ε, για όλους τους ε, στόχους μας εφόσον δεν έχουμε επιτύχει το MSY. Οπότε πρέπει να δούμε πού θα καταλήξουμε πέραν αυτού όσον αφορά την ε, ε, εμπλοκή στα πολυ... Ε, πολυετή προγράμματα κοιτάξαμε το χρονοδιάγραμμα άκουσα τι είπε ο κύριος Χάτσον και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί εάν προχωρήσουμε προς δεύτερη ανάγνωση και ξεφύγουμε από το στόχο μας και δεν έχουμε απόφαση μέχρι το τέλος του 2013 δεν θα έχουμε μία νομική βάση και θα γίνει το ίδιο το οποίο έγινε με τα νέα τρόφιμα όλα θα καταρρεύσουν και θα είμαστε στο έλεος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να διατυπώσει μία νέα νομοθετική πρόταση, πράγμα το οποίο ενδέχεται να πάρει μερικά χρόνια ακόμη και μερικό χρόνο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και υπάρχουν πάρα πολλοί ψήφιροι ότι ε, εφόσον υπάρχει το θέμα της περιφερειοποίησης ορισμένοι ε, επίτροποι θα ήθελαν να ε, ξεφύγει το χρονοδιάγραμμα και λέγουν ότι εάν υπάρχει ε, μία ε, ρύθμιση περιφερειοποίησης για την κοινή αλευτική πολιτική. Το ίδιο θα γίνει μετά και για την κοινή γεωργική πολιτική. Οπότε προσέξτε, μην ε, βοηθήσετε τους αυτούς οι οποίοι θέλουν κάτι τέτοιο αντί να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κατευθείαν. Ευχαριστώ. θέλω να σας πω ότι ε, το να επιτύχουμε την ε, ε, κοινή πολιτική και τα αποθέματα είναι κάτι το οποίο έχουμε δεχθεί και ε, τα περισσότερα κράτη έχουν συμφωνήσει ε, σε αυτό στο Johannesburg για την βιώσιμη ανάπτυξη το 2002 αλλά υπήρξε στη συνέχεια και φέτος το καλοκαίρι στο Ρίο Janeiro μία νέα διεθνής διάσκεψη και επί του ιδίου θέματος και όλοι ζητούν και κάνουν έκκληση επιγόντως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Οπότε ενώ το 2000 δύο είχαν ζητήσει έναν στόχο, δεν είναι δυνατόν το 2012 να επανέρχονται και να λέγουν ότι εμείς οι πλούσιες χώρες δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη μεγίστη βιώσιμη απόδοση σκέφτονται μάλλον τις υποανάπτυξη χώρες και είναι ντροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή να μην μπορέσει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει από το 1994 έχει διακηρύξει και επιβεβαιώσει σε διάφορες διεθνείς διασκέψεις ε, και επανήλθε σε αυτές στο Ρίο προλίγων μηνών. Ε, για την περιφερειακή ανάπτυξη αυτό σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό σε ορισμένες χώρες από ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ισπανία η οποία λέγουν δεν μπορούμε να το πράξουμε μπορούμε να το υλοποιήσουμε και πρέπει να το αποδείξουμε σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Πένας τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Επιτροπή σας για το εύρος των ε, τροπολογιών, το πλήθος τους, αλλά και την δημιουργικότητα που τις υπαγόρευσε. Θα κάνω μια γενική εκτίμηση εγώ και μετά θα σας ε, γίνει από τον συνάδελφο και η εκτίμηση των συμβαστικών τροπολογιών όταν έρθει η ώρα, αλλά θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε μια επικοδομητική στάση. Στόχο στόχος μας είναι σαφής. Είμαστε ω Επιτροπή ευέλικτοι ω δε προς τις πρακτικές λύσεις που θα επιτρέψουν ε, την ε, θέση την υλοποίηση των στόχων μας. Είμαστε επίσης ευέλικτοι. Μια θετική στάση λοιπόν έναντι αυτών των τροπολογιών. Και αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω τους στόχους που καθοδηγούν την Επιτροπή στην εξέταση των τροπολογιών αυτών και βέβαια και στο μέλλον σε σχέση με τις συμβαστικές τροπολογίες για την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι γνωστές οι θέσεις μας. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω τις πρόσφατες πρακτικές, ε, την εμπειρία μας καλύτερα από την πρακτική, που αποδεικνύει ότι Ε, αλλιευτικά αποθέματα τα οποία είχαν και υπεραλλιευθεί στο παρελθόν, ύστερα από ένα χρονικό διάστημα και την εισαγωγή κατάλληλων μέτρων, αποκαθίστανται. Υπάρχουν δηλαδή επιτυχίες σημαντικές και μπορούμε να δούμε, να διαγνώσουμε ακόμη και οικονομικά συμφέρουσες εξελίξεις. Άρα έχει αποδειχθεί η αξία αυτών των μέτρων που αποσκοπούν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα, εάν θα δούμε χάρη στις ε, ε, επιλογές αυτές οικονομική απόδοση ε, με, τις, με την αποκατάσταση των αλλιευμάτων μας, αυτό θα έρθει μετά. Δηλαδή πρώτα θα γίνει η αποκατάσταση των αλλιευμάτων και μετά θα έρθει και η οικονομική απόδοση. Ξέρω ότι αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση των αλλιευμάτων και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί βαίνουν προς τον ορθό δρόμο. Με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι υπάρχει συνειδητοποίηση σαφής ε, ε, από πλευράς της Επιτροπής σας για το θέμα αυτό και είναι για την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα σημαντικό να ε, τηρηθεί η κύρια προτεραιότητα, δηλαδή να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το εξειδικευμένο αυτό χρονοδιάγραμμα για της, ε, για την ε, αλία στην Ευρώπη, για τις μεταρρυθμίσεις, μέσα στους στόχους και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί. Για να επιτευχθούν οι στόχοι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει και το επαναλαμβάνω, ότι είμαστε ευέλικτοι και με θετικό πνεύμα δεχόμαστε και εξετάζουμε τις τροπολογίες που θα κατατεθούν. Για το πολιετές σχέδιο τώρα Πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι ότι πρόκειται για το κατεξοχήν μέσον διαχείρισης της αλίας των ελευμάτων. Άκουσα τις ε, ε, επόψεις και προτάσεις ε, των πάντων με ιδιαίτερη προσοχή. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και με το Συμβούλιο για την διαχείριση και τις αρμοδιότητες στη διαχείριση μέσα στο πολίτες σχέδιο και βέβαια η Επιτροπή σας ε, διαβεβαιεί για κάθε διάθεση υποστήριξης, ε, βοήθειας, αρρωγής προς το Κοινοβούλιο, οτιδήποτε χρειάζεστε για να ε, προχωρήσετε στη δουλειά σας και βέβαια να καταλήξουμε όλοι μαζί σε μια ικανοποιητική λύση. Για την περιφερειοποίηση τώρα, η αποκέντρωση και για να απαντήσω στα όσα είπε ο Στίβενσον. Η Επιτροπή έχει εξηγήσει ήδη και επαναλάβει ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει μέχρι το βαθμό που επιτρέπει ως προς την αποκέντρωση, την περιφερειοποίηση, η συνθήκη της Λισαβόνας. Το όριο είναι αυτό που χαράσει η συνθήκη της Λισαβόνας. Όσον αφορά τη Συμφωνία Γενικών Προσανατολισμών του τελευταίου του Συμβουλίου, του Ιουλίου δηλαδή, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι την κύρια δυσκολία, τα κύρια προσκόμματα δεν θα τα δείτε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αρκεί να διαβάσει κανεί τι γενικέ κατευθύνσει του Συμβουλίου και θα καταλάβει τι εννοώ. Άρα η Επιτροπή δεν προσπαθεί να εμποδίσει τις εξελίξεις. Τουναντίον είμαστε ευέλικτοι, κοιτούμε και εξετάζουμε κάθε λύση με μία μόνο ουσιαστικά προϋπόθεση, δηλαδή την τήρηση, αυστηρή τήρηση των όρων της συνθήκης της Λισαβόνας όπως είναι αυτονόητο. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις τροπολογίες, πολύ άριθμες όπως έχουν κατατεθεί, αλλά υπενθυμίζουμε ταυτόχρονα ότι δεν πρέπει να λησμονούμε πως βρισκόμαστε, και πρόκειται εδώ για αλλία για ε, κοινέ αρμοδιότητες μαζί με τα κράτη-μέλη και έτσι ταυτόχρονα δεν πρέπει να επισημάνω ότι έχουν αποδείξει και πολλές μελέτες στα θέματα των ε, ηχθειοκαλλιεργειών ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τις αρμοδιότητες που έχουν, παραδείγματα της εκχωρής αδειών, εκμετάλλευσης κ.ο.κ. Άρα οτιδήποτε κάνουμε στον τομέα της ηχθειοκαλλιέργειας είναι καταδικασμένο σε αποτυχία εάν δεν συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, εάν και τα ίδια δεν στρατευτούν στον ίδιο δρόμο. Και έτσι για λόγους και στρατηγικούς καλό θα είναι να αποφύγουμε τις ε, δυσκολίες αυτές που προκύπτουν στο εθνικό επίπεδο. Αυτά κύριε Πρόεδρε εν ολίγης και σε αδρές γραμμές ε, τα όσα μας καθοδηγούν στον δρόμο μας ε, στην πορεία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρόντους τώρα για να ολοκληρώσουμε. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι κατέστη σαφές τη σπάση και από τη συζήτηση που μόλις ε, διεξήχθη ότι όλοι συμφωνούν ότι όλοι επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, εν τέλει δηλαδή ένα καλό αποτέλεσμα. Θα επιδιώξω τώρα να ε, τοποθετηθώ στις διάφορες ε, προτάσεις που ακούστηκαν, καταρχάς της κυρίας Φράγα. Κυρία Φράγα, από τις τροπολογίες σας πολλές είναι αυτές τις οποίες διάβασα με θετικό πνεύμα και που με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι να να μην αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα μεταξύ μας. Αλλά τώρα το να περιμένουμε ότι μετά τις 20 Ιουλίου και μέχρι τώρα όλες οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατευθεί θα είναι έτοιμες και μεταφρασμένες στην κάθε γλώσσα είναι νομίζω ε, αδύνατον, ε, απρο, ε, απρόσμενο και είναι και δύσκολο να περιμένει κανείς ότι θα υπάρχουν και οι συμβαστικές τροπολογίες έτοιμες. Πάντως προσπαθούμε να προχωρήσουμε βήμα το βήμα, αυτό το έχω πει και από πριν σε τελευταία ανάλυση και έχει νόημα μόνο όταν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα θέματα, όλα τα ζητήματα και όταν έχει κανείς τη γενική εικόνα μπορώ να έχω εγώ και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε σοβαρές δυσκολίες και διαφωνίες να μπορέσουμε τροπολογίες οι οποίες μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους, είναι τόσο συγγενείς διατύπωσή τους και μπορεί να διαφέρει μόνο μία μικρή λέξη, να τις ενοποιήσουμε μέσα σε μια συμβαστική. Βεβαίως τα σημεία της καμπής θα είναι αυτά που αφορούν την μεταρρύθμιση, την ουσιαστική μεταρρύθμιση και βεβαίως εγώ δεν θέλω να προχωρήσω κατά τρόπον εριστικό ή πιεστικό στη μεταρρύθμιση αυτή. Με τελευταία που θα ήθελε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στο δυνατόν πιο απρόσκοπτα σε μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση. Και θα κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Ταυτόχρονα, ωστόσο, όμω, δεν μπορώ και να απαιτήσω περισσότερα από του συνεργάτε μου και τι συνεργάτηδέ μου από ό,τι κάνουν ήδη. Μέχρι αργά το βράδυ δουλεύουν μαζί μου. Από μένα περιμένετε όσα θέλετε. Απαιτήστε περισσότερα από μένα. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ προφανώ και θα παραιτηθώ από τι διακοπέ μου, αλλά δεν μπορώ να ζητήσω από τον συνεργάτη μου ή τη συνεργάτη μου να μην πάει διακοπέ για αυτό το λόγο. Έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα και από την ομάδα μου και από τη γραμματεία μου, αλλά και από το δικό μου το προσωπικό, του δικού μου γραφείου, που δουλεύουν μερόνυχτα μόνο γι' αυτό, μόνο για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τι συμβαστικέ τροπολογίε και τη διατύπωσή του. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ, αντιληφθείτε κι εσεί ότι είναι ε, ε, ανθρωπίνω αδύνατον 12 Σεπτεμβρίου να είναι τα πάντα έτοιμα και ολοκληρωμένα στο τραπέζι των συζητήσεων. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα δουλέψουμε από τι 12 Σεπτεμβρίου με βάση όσα έχουμε στη θέση μα. Αυτά λοιπόν και αυτή είναι η έκκλησή μου για κατανόηση. Επίσης ε, για του επιμέρους τομείς πολιτικής, για την αποκέντρωση και όλα τα ζητήματα, βεβαίως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα τα συζητήσουμε όλα όπως πρέπει. Δεν θα μπω όμως τώρα στις λεπτομέρειες. Είναι πολλές οι προτάσεις. Είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις καλές. Εγώ προσωπικώς και νομίζω ότι και οι λοιποί συνάδελφοι έχουν ε, την ίδια αντίληψη ή οι περισσότεροι ε, τουλάχιστον θεωρώ ότι ήταν ε, μάλλον αντιπαραγωγική η συνεδρία του Συμβουλίου του Ιουλίου διότι βλέπουμε ότι υπήρξε αντιγραφή ουσιαστικά των κειμένων του Συμβουλίου, των προηγουμένων κειμένων και ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αντιληφθεί το Συμβούλιο ότι και εμείς εδώ έχουμε την δυνατότητα και την ευφυΐα να διατυπώνουμε τις δικές μας προτάσεις, να σχηματίζουμε τις ιδέες μας και ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλαμβάνουμε λέξη προς λέξη τα όσα έχει προτείνει το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να είμαστε κάπως πιο επιφυλακτικοί και να περιμένει και το Συμβούλιο από πλευρά του να δει τι θα ετοιμάσει το Κοινοβούλιο για τον κύριο Φεραίρο, ο οποίο θεωρεί ότι ήδη έχουν κλείσει όλα τα θέματα. Α, έφυγε, δεν είναι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η διατύπωση θα πολύ σκληρή όπω την ε, χρησιμοποίησε. Ε, ότι θεωρεί ότι τα έχει κλείσει όλα τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί απλώ τα επαναλαμβάνουμε. Θα του έλεγα λοιπόν, αν ήταν εδώ, ότι δυόμιση χρόνια δουλεύουμε μαζί, εντατικά συνεργαζόμαστε και νομίζω ότι έχει καταστεί σαφέ για του πάντε ότι είμαστε σε θέση όταν χρειάζεται να στραφούμε, να αντισταθούμε καλύτερα στις θέσεις και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Έχουμε τις δικές μας θέσεις και έχουμε βέβαια και το μεγάλο όπλο της συναπόφασης, το οποίο πιστεύω μπορούμε να αξιοποιήσουμε. για τον κύριο Ντέιβις. Είπε ο κύριος Ντέιβις, όπως και η κυρία Λουβίν, ότι... Πολλά πράγματα ακόμη μπορούν ε, να συζητηθούν περαιτέρω και σε σχέση με το ε, Συμβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν πήγα στην ε, Γερμανική ημέρα της Αλίας, ένα μεγάλο συνέδριο, δόθηκε η εντύπωση από μου δόθηκε η εντύπωση από τα όσα άκουξα ότι το Συμβούλιο έχει κλείσει όλα τα θέματα και τα αποφασίζει μόνο του. Ε, όχι λοιπόν, αυτό δεν θα το δεχθούμε και θα πρέπει να καταστήσουμε σε θέση το Συμβούλιο ότι και εμεί είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δουλειά μα σωστά και επικοδομητικά. Και ε, θα ήθελα να ευχαριστώ τον Στιούαν για την ε, τοποθέτησή του. Νομίζω δεν μπορούσε να είναι πιο εύγλωτος. Βεβαίως και έχουμε υποχρέωση να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας και να τηρήσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε αυτό. το να πιστεύει κανεί ότι μπορούμε να δουλεύουμε μέχρι το 2014-2015 στο θέμα αυτό προφανώ δεν είναι σοβαρό. Και βεβαίω πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Είχα και εγώ καταθέσει μια πρόταση η οποία θα πήγαινε μέχρι τις αρχές της των θερινών διακοπών για την επεξεργασία όλων των τροπολογιών με τη, με, τη μετάφρασή τους. Μετά μου ζητήθηκε να παρατείνω και εγώ την προθεσμία μου και ε, το δέχτηκα. Ε, και τώρα θα πρέπει να παρατείνουμε λίγο τις προθεσμίες στο βαθμό που είναι δυνατόν, διότι ξέρω ότι με όλες τις προσπάθειες που κάνω χρειάζεται να πιεστώ πολύ για το χρονοδιάγραμμα. Και παρακαλώ όλες και όλους ε, τους συναδέλφους, ε, γιατί όλοι έχουμε την υποχρέωσή μας, όχι μόνο για το Κοινοβούλιο, αλλά έχουμε υποχρέωση απέναντι στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κάνουμε μια προσπάθεια παραπάνω, ας ξενυχτήσουμε μια βραδιά, ας κάνουμε την προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά εφέτος για να περάσει στην Ολομέλεια και να κλείσει το θέμα από πλευρά μας. Είμαι πεπισμένη ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και είμαι πεπισμένη ότι αυτός είναι ο στόχος που θα επιτύχουμε πραγματικά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία, έστω αν όχι συνένεση, η οποία θα ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό όλους τους συναδέλφους. Έχουμε δουλειά ακόμη πολύ και πάλι επαναλαμβάνω ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και περιμένω περαιτέρω συνεργασία και προσεχή συνεδριάζεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κλείνει το θέμα αυτό και έτσι περνάμε στο επόμενο με τη συμφωνία σας. Γνώμη που αφορά την τροπή του κανονισμου αριθμό αριθμός 2371-2002, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας ζήτησε να εργαστούμε με προσοχή και επιμέλεια, όπως άλλωστε πράξει ο κύριος Χάτσον, ο εισηγητής μας, τον οποίο και συγχαίρω, συγχαίρω και για τα πολύ ταχεία δουλειά του, του δίνω το λόγο να μας κάνει την παρουσίαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας ε, εκπλήξει φαντάζομαι το γεγονός ότι η Κομισιόν τελικά ε, αναγνώρισε στην ε, παρουσίαση αυτής της, αυτού του κανονισμού είναι ότι το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται είναι πολύ ζωρισμένο. Εν πάση περιπτώσει, η πρόταση αφορά την επέκταση του χρονικού ορίου σε σχέση με το ισχυρό καθεστώς πρόσβασης των 12 μιλίων για δύο ακόμα χρόνια. Ε, ήμουν ιδιαίτερος επικριτικός, όπως το ξέρετε όλοι, όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική. Δεν είναι πολλά τα σημεία της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, για τα οποία θα μπορούσα να μιλήσω με καλά λόγια. Είμαι πολλά χρόνια βουλευτής και πολύ σπάνια συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό τώρα πραγματικά με σοκάρει το γεγονός ότι θα συμφωνήσω με αυτά που λέει. Όταν λέει ας πούμε ε, στο, στην Πράσινη Βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχολιάζει ότι έχει γενικά λειτουργήσει ικανοποιητικά και μπορεί ακόμα και να ενισχυθεί το καθεστώς των ζωνών των 12 μιλίων, ε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Ε, επίσης, σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι το καθεστώς είναι πολύ σταθερό και τα αποτελέσματά του είναι σταθερά ικανοποιητικά. Ε, η αρχή, λοιπόν, ε, είναι καλή, αναγνωρίζεται η επιτυχημένη ε, αρχή αυτή και ε, επομένως ε, θεωρώ ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την, τα δικαιώματα τους όσον αφορά αυτήν τη διαχείριση της ζώνης των 12 μιλίων γιατί τα αποτελέσματα είναι καλά. Πρέπει να σας πω ότι ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα να προτείνω στα πλαίσια αυτής της ε, ε, έκθεσης ε, να γίνει μόνιμη αυτή η διαδικασία. Επίσης, αισθάνθηκα μεγάλη πρόκληση του να υποβάλω τροπολογίες έτσι ώστε τα 12 μίλια να γίνουν ακόμα περισσότερο, να μεγαλέσει περισσότερο η παράκτια ε, ζώνη, ε, κάτι που είχα προσπαθήσει να κάνω και στην προηγούμενη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής. Εν πάση περιπτώσει, κατάλαβα στο τελικά ότι αυτή η συγκεκριμένη έκθεση δεν είναι το κατάλληλο μέρος ε, για να προτείνουμε κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να ενταχθεί στη γενικότερη συζήτηση της μεταρρυθμιστικής δέσμης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Επομένως, πέρα από τα όσα σας είπα ήδη, ε, σας λέγω ότι πρέπει να δεχτούμε την πρόταση της Επιτροπής το, 12, το καθεστώς των 12 μιλίων θα πρέπει να παραταθεί ε, για δύο τουλάχιστον ακόμα χρόνια επί τη βάση των όσων ε, είπα προηγουμένως και όσον αφορά τώρα ε, το γενικότερο πλαίσιο σχετικά με την καθιέρωση SAE αυτού του, προγρατού θέματος θα συζητηθεί σε άλλα φορά. Η κυρία Φράγα έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Φερέιρα μετά. Ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Συγχαίρω τον κύριο Χάκτον ε, για την εργασία του και βεβαίως θα πω ότι για μία ακόμα φορά συμφωνώ με τα συμπεράσματά του. Συμφωνώ ε, με το σημείο 1, σημείο 1 για, και καθώς επίσης και με το σημείο, το σημείο 4 όλα αυτά θα πρέπει ε, να ε, δυναμωθούν. Ε, επίσης, εάν γίνουν προτάσεις για ουσιαστικές τροποποιήσεις της ελευθερικής πολιτικής, θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια της εκθέσεως ρόντου και όχι εδώ. Εδώ υπάρχει μία ε, αρχή η οποία πρέπει να εφαρμόζεται και νομίζω ότι υπάρχει γενικευμένη συμφωνία σχετικά με τα 12 ε, μίλια και θα πρέπει να ε, κρατηθούμε σε αυτά τα 12 μίλια και να μην διευρύνουμε είτε τα μίλια είτε την συμφωνία. Υπάρχει ήδη, υφίσταται ήδη συμφωνία και επομένως δεν συμφωνώ αυτή η παρέκκληση να γίνει ε, μόνιμη ε, και ούτε συμφωνώ να ξεπεραστούν τα 12 μίλια, γιατί ούτως ή άλλως αυτό αντιτίθεται στην αρχή της ελεύθερης πρόσβασης ε, που, που μας είναι για πολλούς μεταξύ ημών ιδιαίτερος προσφυλής. Κατά τα λοιπά δεν έχω κάτι εναντίον της εκθέσεως αυτής. Οπωσδήποτε θα συμφωνώ και εγώ με την διετή παράταση όπως το προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ε, όπως προβλέπεται στον βασικό κανονισμό. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάκτον για την ε, εργασία την οποία έχει κάνει. Αντίθετα από την ε, κυρία Φράγκα, εγώ θα, ε, θα ήθελα να συμφωνήσω πλήρως με την ε, πρότασή του. νομίζω ότι θα πρέπει βεβαίως να θεωρήσουμε την την μονιμοποίηση αυτού του μέτρου, ε, όχι εδώ, αλλά στα πλαίσια της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, θα συμφωνήσω επίσης για όλα, με όλα όσα είπε ο κύριος Χάκτον όσον αφορά την διαχείριση αυτών των ζωνών των 12 μιλίων. Δεν θα συμφωνήσω με την κυρία Φράγα. Νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν δεκτές και όπως και ο κύριος τον είπε πολλά πράγματα πάνε κακά, άσχημα με την κοινή ελευτική πολιτική, αλλά υπάρχει ένα το οποίο λειτουργήσε καλά. Είναι αυτό το μέτρο της ειδική διαχείρισης της ζώνης των 12 μιλίων. Ε, και από τη στιγμή που ένα ε, μέτρο πάει καλά, νομίζω ότι αφενός είναι απαραίτητο να το διατηρήσουμε, αφετέρου είναι ορθό να το διευρύνουμε. Επομένως, Πιστεύω ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και βεβαίω θα πρέπει να είναι δυνατόν να περάσουμε και πέρα από τα 12 μίλια, ξεπερνώντα λοιπόν και το όριο της υφαλοκρηπίδα, εάν ε, αυτό είναι ε, ε, δυνατόν. Σε περιοχές όπως είναι, σε περιπτώσεις όπως είναι ας πούμε τα νησιά, θα πρέπει να γίνει μια ειδική συζήτηση. Θα μπορούσε να διευρυνθεί η ζώνη των 12 μιλίων στο βαθμό που δεν θίγονται κάποια άλλα ευαίσθητα ε, θέματα και βεβαίως Είναι σαφές ότι με την επέκταση της αποκλειστικής ζώνης οι παράκτιες κοινότητες ε, θα ε, ευνοηθούν, θα, θα, έχουν θετική επίπτωση λοιπόν, θα έχει θετική επίπτωση στις παράκτιες κοινότητες. Ε, είναι γεγονός ότι υπάρχουν και περιοχές στις οποίες θα πρέπει να επιτραπεί η ελευθερία πρόσβασης, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να διευρυνθούν οι αποκλειστικέ ζώνες. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν τα καλά σημεία, το καλό σημείο της κοινή ελευθερικής πολιτικής θα πρέπει ε, να διατηρηθεί, αλλά βεβαίω και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διατηρηθούν τα αλλιευτικά αποθέματα. Συμφωνώ λοιπόν, συμφωνώ απολύτω με όσα είπε ο ε, συνάδελφος ε, Χάκτον ε, και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα θετικό σημείο στην αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να το διατηρήσουμε και βεβαίως η αποκίνδυνοση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής δεν είναι καθόλου κακό πράγμα. Επομένως, Περιμένω, περιμένω τις εξελίξεις και όσον αφορά την έκθεση Ρόντουστ, όπου θα, μπορεί να, θα μπορέσει να γίνει μια πολύ καλή συζήτηση και ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουμε τελικά να συμφωνήσουμε με την επέκταση της αποκλειστικής ζώνης, οποτεδήποτε και οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Um, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ο Στιούαρτ Στίβενσον και προηγουμένως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η δονιστές, ξεκίνησαν ορισμένες συζητήσεις για τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο και να ε, διαπραγματευτούμε σοβαρά για τα μακροπρόθεσμα προγράμματα και να εντοπίσουμε ορισμένες εκθέσεις που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν για να ενοχληθεί το Συμβούλιο συμφωνώντας με όλες τις πολιτικές ομάδες. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι ναι μεν πρέπει να επεκτείνουμε τα ισχύοντα περιθώρια, όσον αφορά όμως το χρονοδιάγραμμα δεν είμαι τόσο βέβαιος. Μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε ότι ε, θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του συζητήσεων του Συμβουλίου κάθε τρίμηνο μέχρι ότου το υιοθετήσουν θα ήταν μια καλή ιδέα, αλλά η επιφύλαξή μου εδώ είναι ότι ναι μεν χρειάζεται να επεκτείνουμε την ισχύουσα νομοθεσία αλλά ίσως θα πρέπει να γίνει για τρεις μήνες ή έξι μήνες και όχι για δύο χρόνια και πέρα διότι αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα, ορισμένες δυσκολίες σε ορισμένους ψηφοφόρους μας και στο Συμβούλιο το οποίο αντιτίθεται και ως εκ τούτου είναι ένα σοβαρό εργαλείο. Αλλά αυτή είναι η επιφύλαξη που έχω στις ε, παρατηρήσεις που άκουσα μέχρι τώρα. Η κυρία Κούπερ τώρα, για την ευρωπαϊκή ο κύριος Κούπερ για ε, ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να συγχαρούμε τον εισηγητή. Είναι καλό να βλέπουμε μία έκθεση η οποία υιοθετεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι και στα συμπεράσματα και ε, ουσιαστικά τα δύο θέματα όπου ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, δράσει είναι θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επισέλθω τώρα σε λεπτομέρειες ε, αλλά ε, νομίζω ότι προχωρούμε στην έγκαιρη υιοθέτηση της πρότασης και δεν είναι κακό αυτό. Ευχαριστώ ο εισηγητής για να κλείσει. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Απαντώντας στην κυρία Φράγκα, ίσως δεν θα εκπλαγεί, δεν θα έπρεπε να εκλαγώ εγώ ότι δεν δέχεται δύο-τρία από τα συμπεράσματά μου, αλλά ίσως υπάρχει παρανόηση, διότι δεν λέμε εδώ ότι πρέπει να επεκταθεί ΕΣΑΗ, e, αλλά απλώ ότι πρέπει να υπάρξει μία επέκταση. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι λογικό να ζητάτε, τουλάχιστον να εξεταστεί κατά τρόπον ώστε να μην συνεχίσουμε όπως πάμε τώρα. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο ε, ουσιαστικά Έχουμε το μόνο σημείο της κοινή ε, ε, αλευτικής πολιτικής ε, το επί του οποίου θα έπρεπε να συζητήσουμε σχετικά με τις αρχές της δίκαιης και ίσης πρόσβασης κατά τρόπον ώστε να σταματήσουν οι καταστροφικές ε, ε, ροές ε, της τωρινής κατάστασης και να ζητήσουμε να διατηρηθεί το Καθεστώ των 12 μιλίων διότι έτσι ε, θα αποφύγουμε αυτά τα οποία γίνονται τώρα και θα μπορέσουμε τουλάχιστον να βελτιώσουμε το σύστημα. Νομίζω όμως ότι έχουμε μία ευκαιρία η οποία δίνεται για μία αναθεώρηση της πολιτικής και ελπίζω ότι οι ευρωβουλευτές θα συμφωνήσουν διότι νομίζω ότι ουσιαστικά πρέπει να υπενθυμίσουμε ορισμένα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός είναι ο στόχος μας ότι πρέπει να διατηρήσουμε το όριο των 12 μιλίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τα θέματα που τίθενται στο σημείο 2 και 3 απλούστατα θα πρέπει να κοιτάξουμε να αποδεχθούμε ε, ορισμένα θέματα για να μπορέσει να συνεχίσει η συζήτηση. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ε, πω ότι ε, η προθεσμία για τις τροπολογίες έχει καθοριστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα στο 9 αλλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται για τη Συμφωνία Αλλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως αφενός, της κυβέρνησης Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γρυλανδίας. Συζητήθηκε ήδη το θέμα τον Ιούλιο, το Συμβούλιο θα το συζητήσει 18 ε, ενάτου το πρωτόκολλο θα υπογραφεί ε, ο πρωτόκολλο συμφωνίας όπως είπα θα ε, υπογραφτεί στις 18 Ενάτου και ο εισηγητής παρουσιάζει τώρα το σχέδιο της εκθέσεώς του. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Γρυλανδίας ανέρχεται σε πολλά χρόνια και θεωρείται ένα βασικό στοιχείο συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Βορρά για την εκμετάλλευση των πόρων. Το, ε, το αποτέλεσμα που επετεύθη ήταν θετικό και ε, η έρευνα, η επιμόρφωση του προσωπικού συνέβαλε στη βιωσιμότητα της αλίας στη Γρυλανδία. Το νέο πρωτόκολλο προβλέπει ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει με 85 εκατομμύρια κάθε χρόνο για να μπορέσει να στηρίξει τον τομέα της αλληλείας της Γρυλανδίας. Με το νέο όμως πρωτόκολλο η κοινή επιτροπή τώρα θα αποφασίσει ποιες θα είναι οι αλληλευτικές ευκαιρίες κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί εις ε, τις ανάγκες της βιομηχανίας και να συμβάλλει στη διατήρηση της αλληλείας στο σημείο αυτό. Η βιώσιμη αλληλεία είναι ένα θέμα που θα πρέπει να προωθηθεί ε, ε, γιατί μέχρι στιγμής η αρχή αυτή συνέβαλε εις την ευημερία και των δύο ενδιαφερομένων και έχει ε, γίνει εξέταση των ε, επιστημονικών πτυχών και των τεχνικών θεμάτων πρώτης καταρτήσεως του νέου πρωτοκόλου ε, και τα μέτρα στηρίξεως για την περιοχή ιδίως σε σχέση με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα είναι αποδοτική μακροπρόθεσμα και θα πρέπει ε, να εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω λοιπόν να δοθεί η ευκαιρία να υπάρξει μία πιο στενή παρακολούθηση του πολιετούς προγράμματος και επιπλέον εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν παρατηρητές να μπορέσουν να συμμετέχουν στις τις διεργασίες της ε, κοινή ε, ε, Επιτροπής Διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ και προτείνω να υιοθετηθεί το πρωτόκολλο αυτό. Ευχαριστώ τον κύριο Κρίστενσεν για την εκτενή του έκθεση σαν εισηγητή και συμφωνούμε ακριβώς όπως το παρουσίασε ε, η Επιτροπή ε, οικονομικών επίσης ε, έχει υιοθετήσει αυτό το θέμα αλλά θέλω να κάνω μία ερώτηση. Οι δυνατότητες της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά τη χρηματοδότηση και οι αποζημιώσεις οι οποίες καταβάλλονται για την ευρωπαϊκή πολιτική αλληλείας ελπίζω ότι θα υιοθετηθούν διότι 22.000 τόνοι ψάρια φτάνουν από την ε, Γρυλανδία κάθε χρόνο και συνολικά έχουμε 32.000 τόνους Οπότε ε, αυτό συνάδει με ε, τους, τις διατάξεις για την εξοικονόμηση πόρων. Βέβαια δεν ξέρω ε, πόσα εκατομμύρια ευρώ είχαμε συμφωνήσει στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Τώρα μιλάμε για 17,8 και υποθέτω ότι έχουν σωστά συμπεριληφθεί όλα τα στοιχεία σχετικά με τους 30.000 τόνους. Θέλω να ξέρω αν αυτές οι πληρωμές γίνονται κατευθείαν προς τη Γρυλανδία και να ξέρω τι ε, δυνατότητες έχουμε για τη Γρυλανδία ε, διότι πλέον η Γρυλανδία δεν ελέγχεται όσον αφορά την αλληλευτική εποπτεία από την κυβέρνηση της Δανίας ενός κράτους μέλους αλλά από άλλο οργανισμό και ως εκ τούτου θα πρέπει ε, να έχουμε εξ αυτών και τις τις ε, εκθέσεις και ε, τις τεκμηριώσεις των στοιχείων. Αυτή είναι η απέτησή μου, κατά τα άλλα συμφωνώ. Η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το κείμενό του. Μου φαίνεται καλό, ισορροπημένο. Θα ήθελα ξεκινώντα να κάνω μια γενική παρατήρηση και στη συνέχεια θα διατυπώσω ερωτήσεις. Στην περίπτωση της Γρυλανδίας, Έχουμε πολύ συγκεκριμένη συμφωνία, όπως άλλωστε συμβαίνει όπως άλλωστε δεν συμβαίνει με το Μαρόκο, την Γουινέα, Μπισάο και άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι στην περίπτωση της ανανέωσης του πρωτοκόλου διατηρούνται οι διαφορές που είχαμε πάλι σε σχέση με τις λοιπές και ειδικέ ε, συμφωνίες. Η μία διαφορά είναι ε, αυτή που έχει να κάνει με την κατανομή των ποσοστώσεων, που πάλι είναι διαφορετική και βλέπουμε ότι οι χώρες πλειοδότες αποφασίζουν, ενώ στις άλλες ε, συμφωνίες βλέπουμε ότι αν ένα συγκεκριμένο στόλος δεν αξιοποιεί τις αλληλευτικές ποσοστώσεις, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για να τις αναδιανύμει. Αυτή η διαφορά λοιπόν συνεχίζεται. Εγώ θεωρούσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να ενοποιήσει τις ειδικέ συμφωνίες για το πράτη. Ε, κάτι άλλο. που έχει να κάνει με τους πλειοκτήτες, οι οποίοι στις ε, ε, Μαυριτανίας πληρώνουν έως το 40%. Ο εισηγητής λέει επισημαίνει, όπως και στην έκθεση αξιολόγηση, ότι στο προηγούμενο πρωτόκολλο ήταν 15-85% ε, η κατανομή. Εάν όμως παραμείνουν αυτά τα τέλη και δεν τροποποιηθούν όπως έχει γίνει αλλού, παραμένει η διαφορά και μάλιστα αυξάνεται. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή σε διαφορά σε Αναλογία 10 προς 90. Γιατί λοιπόν ε, μόνο 10% πλειοκτήτης ενώ στην περίπτωση της ε, Μαυρετανίας είχαμε φτάσει στο 40% και γιατί αυτό το ρωτώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί διαφυλάσσεται αυτή την ε, απόκληση. Και όταν μας λέτε ότι θα πρέπει να πληρώνουν πάντα περισσότερα οι πλειοκτήτες, γιατί ε, εδώ να υποχωρούμε και να ζητούμε κάτι τόσο πιο περιορισμένο. Κάτι ακόμα. Στον ε, κάβουρα του χιονιού, όπως ονομάζεται, ερωτώ, ή τον πολικό κάβουρα, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Έχετε μια αλληλευτική δυνατότητα ε, παραδοσιακή, που όμως δεν αξιοποιήθηκε ποτέ, διότι η Γρυλανδία που έχει τις αλληλευτικές δυνατότητες όταν ανοίγει η αλληλευτική περίοδος κλείνει την πρόσβαση στο αλίευμα. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στην έκθεση. Η μόνη περίπτωση ε, για τον κάβολα της Αρκτικής είναι αυτή που αφορά μια εταιρεία συγκεκριμένη που έχει ειδική συμφωνία με την Γρυλανδία και ε, δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τις συμφωνίες με την ε, για τον ε, κάβουρα της Αρκτικής ενώ δεν μας αφορά πλέον. Δεν έχουμε ποτέ λιεύσει κάβουρα της Αρκτικής και το μόνο καράβι που ενδιαφερόταν τώρα έχει ειδική συμφωνία και δεν εντάσσεται σε αυτήν της Γρυλανδίας. Επομένως, ε, ποιος ο λόγος. Άλλη ερώτηση. Παραδοσιακή. Μας λέτε ότι τα Ε, σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καταβάλουν, θα πρέπει να ε, ζητούν μια επιπλέον ποσότητα και να καταβάλουν ε, το σχετικό τέλος για την ποσόστοση, την επιπλέον ποσόσταση που ενδεχομένως όμως να μην χρησιμοποιήσουν. Γιατί λοιπόν να πληρώνουν τα καράβια μας για ποσοστώσεις αλληλευτικές που δεν αξιοποιούν, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει. Και πρέπει να πω ότι την ερώτηση αυτή έχω ξανακαταθέσει αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λόιβεν, και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Βλέπω ότι ε, λειτουργεί ικανοποιητικά, αρκετά ικανοποιητικά αυτή η συμφωνία βεβαίω παρουσιάζει σε πολλά επίπεδα απλών ανακτήματα για την Κρυλανδία. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. υπάρχουν ενδείξεις ότι ο γάδος ε, και άλλα είδη χθείων, όπως λέει και ο εισηγητής, μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο, γιατί κοίταξα το σχετικό site, τη σχετική του σελίδα, ε, δεν αφορά μόνο αυτά τα είδη, γιατί αναφέρεται ο γάδος μένα στην ε, περιοχή 1, Αλλά επίσης βλέπουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχει πρόταση από την ίσες ISIS για μηδενική ποσόστοση και διαφοροποίηση η οποία τελικά οδηγεί σε σύγχυση για παράκτιο γάδο ή ανοιχτή θαλάσσης. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καταλάβω πώς βοηθούμε την, τα βιώσιμα, την ανάπτυξη βιώσιμων αποθεμάτων επίσης. βλέπω ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα διαχείρισης για το κοκκινόψαλο της Νορβηγίας. Δεν είναι γνωστά τα αποθέματα. Δεν βλέπω ακριβώς δηλαδή πως είναι δυνατόν αυτό το είδος να περιληφθεί στο πρωτόκολλο και κατά τρόπο βιώσιμο. Για δε τον ε, Χάλιμπατ της ε, Νορβηγίας, πάλι, την υπόγλωσσα δηλαδή, εάν δεν έχουμε στοιχεία για τα αποθέματα που να αποδεικνύουν ότι είναι αντίστοιχα με το BMSY, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις επιλογές ως προς την διαφύλαξη των αποθεμάτων, γιατί πρόκειται για ένα είδο το οποίο ζει πολλά χρόνια, υπάρχουν δηλαδή ε, υπάρχουν δηλαδή ψάρια τα οποία φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και άρα η, αποκατάσταση του, ε, της υπόγλωσσας είναι βραδία. Επίσης, στο είδος που ονομάζεται Grenadier, ε, που δεν ξέρω ακριβώς ε, ποιο είναι, αυτό αναφέρεται έτσι στο κείμενο, ε, είναι ένα είδος που ζει στα βαθαία ύδατα, έχει βραφική ανάπτυξη και αποκατάσταση αποθέματος, άρα θα παρακάσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποιο είναι αυτό το είδος. και να μας δώσει και πιο πολλές εξηγήσει. Ε, μήπως καταλάβουμε πόσο ευάλωτο είναι αυτό το είδος. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καταρχάς επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον εισηγητή Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις. Για τις πληρωμές καταρχάς. Η παρουσίαση, ξέρετε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε την προηγούμενη, στην προηγούμενη συνεδρίαση. Υπενθυμίζω ότι το δημοσιονομικό πακέτο για την Γρυλανδία, για την πρόσβαση αφορά τάσεις και εξελίξεις και ταυτόχρονα σημειώνουμε και το αίτημα της Γρυλανδίας, λαμβάνουμε απόψε το αίτημα της Γρυλανδίας για την ενίσχυση της οικονομικής μας ε, συμβολής. Αυτά λοιπόν προς τα οικονομικά στοιχεία. Για την εξισορρόπηση και τα FPA, τη Συμφωνία Ελευτικής Σύμπραξη έχουμε ήδη με την Νορβηγία, την Ισλανδία, τις νησούς Φερόε αντίστοιχες συμφωνίες. Και άρα λαμβάνονται αυτές υπόψη κατά την επεξεργασία της συμφωνίας που είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις λοιπές χώρες. Ως προς τη συμβολή το τέλος αδειοδότησης. Η Επιτροπή προσπαθεί πάντοτε να ακολουθεί τις αρχές που έχουν οριστεί και μέσα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, δηλαδή δίκαιη κατανομή των τελών, και εδώ πάλι αυτό ορίζεται με βάση την ύπαρξη μη συμφωνιών αλληλευτικής σύμπραξη σε σχέση με την Ορβηγία, Φέρος, Ισλανδία και προσπαθούμε να βρούμε μια καλή ισορροπία ανάλογα με το εάν έχει μια χώρα ή μη τέτοιες συμφωνίες αλληλευτικής σύμπραξης FPA. Για τον Κάβουρα. διατηρήθηκε η κατάσταση όπως έχει για λόγους πολιτικούς έντονης μάλιστα απέτηση χώρας μέλους και δι της Ισπανίας. Ξέρουμε ότι είχαμε και στο παρελθόν ε, ζητήματα. Αφού έδειξε τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον η Ισπανία μέσα σε ένα διαπραγματευτικό πακέτο, το, πακέτο, το ποσόν αυτό διατηρήθηκε. Για τα τεχνικά ζητήματα Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του τρέχοντος πρωτοκόλλου είχαμε αρκετές συζητήσεις με την Ιρλανδία για την επίλυσή τους. Υπενθυμίζω ωστόσο ότι πρόκειται για συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιρλανδίας Δανίας και άρα πρέπει να γίνουν σεβαστοί και οι νόμοι και οι κανονισμοί σχετικοί με την αλληλεία της Γρυλανδίας. Ανάλογα με αυτούς λοιπόν ορίζονται και οι υποχρεώσει. Για την κατάσταση και τις ανησυχίε σχετικέ με τα αλλιεύματα και ιδιαίτερα τα είδη που αναφέρατε. Αν κοιτάξετε το προτινόμενο επίπεδο αποθεματών για το νέο πρωτόκολλο, για τα τρία αυτά είδη που καταγράφονται ως απειλούμενα, το νέο πρωτόκολλο μειώνει σημαντικά τις ποσοστώσεις. Η Επιτροπή προσπαθεί πάντοτε να παρακολουθεί την βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Γι' αυτό ορίζονται κατά αυτόν τον τρόπο το, τα αποθέματα. Για το γάδο τώρα, λεπτομερέστερα. Ίσως να έχετε υπόψη ότι στις συνεδριάσεις μου της Επιτροπής προσπαθούμε πάντοτε να τα συζητούμε, διότι και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια κοινή συμφωνία ελευτική σύμπραξη, γιατί κάθε φορά συζητούμε τι ε, ποσοστώσει για το επόμενο έτο. Και άρα έχουμε θέματα. Αυτέ τι ποσοστώσει, δηλαδή, τι οποίε ε, βλέπετε εδώ, πρέπει να τι δείτε μόνο ω ενδεικτικέ ποσοστώσει. Επίση, τα τελευταία χρόνια και για τον ε, και για τις ποσοστώσεις και για τα προγράμματα διαχείρισης για τη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να σας πω ότι είχαμε συζητήσεις ε, στη συνεδριάση μέχρι τώρα της Επιτροπής και άρα τροποποιήθηκαν κάποια θέματα. Αυτά για τα συγκεκριμένα τρία είδη. Για τα λοιπά, το κοκκινό ψαρο της Νορβηγίας Είχαμε ένα νέο πρόγραμμα διαχείρισης, υιοθετήθηκε πέρυσι και άρα ακολουθούμε ο συμβαλόμενο μέρος τις συστάσεις της ΝΙΑΦΚ. Και έτσι είναι σημαντική η μείωση, διατηρείται ένα ελάχιστο επίπεδο και, και εμείς ακολουθούμε το σχέδιο διαχείρισης του ε, κοκκινού ψάρου της Νορβηγίας. Για το, το υπόγλωσσα της Γρυλανδίας πάλι Προσπαθούμε να διατυπώσουμε μέσα από ένα πρόγραμμα διαχείρισης ε, καλές λύσεις. Ζητούμε από την ε, Γρυλανδία προτάσεις. Και είμαστε λίγο πολύ στα χέρια των παράκτιων κρατών, δηλαδή Γρυλανδία, Νορβηγία και το καθεξής. Ε, ό,τι αποφασίσουν εκείνοι θα πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά έχουμε και στο νέο πρωτόκολλο σε υποσημείωση τις αναφορές των ορίων αλλιεύματος και αλλιευτικής προσπάθειας που θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ετήσιο και το πολυετές ε, πρόγραμμα διαχείρισης. Αυτά τα αναφέρουμε ήδη και όπως είπα πρόκειται για ενδεικτικές ποσοστώσεις που κάθε έτος το Νοέμβριο πριν από την εισαγωγή του κανονισμού ξανασυστούνται στην Επιτροπή. Και πάλι θα πρέπει και εμείς η Επιτροπή ειδικότερα να εξετάσει επιστημονικά στοιχεία και να λάβει υπόψη τις προτάσεις ανάλογα με τις συμβουλές των ειδικών για τον προσδιορισμό των ποσοστώσεων. Επίσης, για τον ε, γρεναδιέρο ή ποντικόψαρο, είχε σημειωθεί ως ε, μια υπολοιματική ποσόστοση. Τώρα τη βλέπετε σε ένα χωριστό πίνακα. Γιατί ήταν ποσόστοση παραλιευμάτων ουσιαστικά. Και έτσι λοιπόν τώρα την ε, ξεχωρίσαμε και τη βλέπετε χωριστά στον πίνακα. Αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με, την, ε, με τις συστήσεις μας και τη συμφωνία μας με την Νορβηγία. Αυτά ως προς προσωστώσεις και νομίζω ότι έχω απαντήσει στις ερωτήσεις ε, στο βαθμό που μπορούσαμε εμείς από πλευράς Επιτροπή, σα ευχαριστώ και πάλι για την έκθεση και για τη συζήτηση. Κυρία Φράγα, ίσως ε, δεν εξεφράστην καλώ γιατί δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματά μου. Εάν δεν κάνω λάθος, εάν δεν κάνω λάθος, ε, και έχω την εντύπωση ότι ε, χάνω λίγο περισσότερο το, το, νήμα με την Επιτροπή. Πάντως, Νομίζω ότι αναφέρθηκε σαφώς ότι πρόθεση ε, είναι να ε, με μια σειρά περίφημων εντό εισαγωγικών συμφωνιών. Η Κομισιόν ε, έχει πει ότι οι πλειοκτήτες θα πρέπει να πληρώνουν όλο και περισσότερα. Ξεκινώντας από αυτό, σε κάθε συμφωνία ο πλειοκτήτης πληρώνει περισσότερο και η Κομισιόν πληρώνει λιγότερο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο κανόνας που εφαρμόζεται ε, σε όλους. Και σας παραπέμπω σε αυτή την περίφημη συμφωνία με τη Μαυρετανία, για να καταλάβετε ακριβώς τι λέω. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση η συμμετοχή ε, των πλειοκτητών είναι όλο και λιγότερη. Ε, ξεκινήσαμε από 15%. Το λέει και ο εισηγητής, το λέει και η έκθεση η αύξηση της οικονομικής αντιστάθμισης είναι μεγαλύτερη, αλλά ε, η συμβολή των ε, πλειοκτητών ε, είναι μικρότερη. Γιατί κάνετε κάτι διαφορετικό από ό,τι έχετε κάνει για τις, στις άλλες συμφωνίες. Νομίζω ότι η ερώτηση είναι σαφής. Για να δούμε, η απάντηση θα είναι εξίσου σαφής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Να σας πω ότι έχουν αυξηθεί ε, τα αλλιεύματα, αλλά ονομαστικά ε, βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα, υπάρχουν και άλλες συμφωνίες οι οποίες ε, βρίσκονται εν ισχύ και οπωσδήποτε αυτή η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με άλλες συμφωνίες το 40% ε, εάν ανταλλάσσετε το 40% ε, βάση αυτών των ε, αλλιεύσεων πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε νέα στοιχεία και για την Ιρλανδία και για άλλες συμφωνίες που έχουμε στην περιοχή οι υποχρεώσεις δεν είναι ίδιες αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω προηγουμένως στην απάντησή μου δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες αδειοδότησης ε, ε, βρήκαμε ότι δεν υπήρχε αντιστοιχεία και συμφωνία με τις ήδη υφιστάμενες συμφωνίες. Κύριε Κρίστανσεν, για να ολοκληρώσετε τη συζήτηση, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα σχόλια αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απήντησε σε ορισμένες από τις τεχνικές ερωτήσεις. Ε, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να απαντήσω, θα είχα δυσκολία να απαντήσω. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός των ε, ψαριών που μπορούν να αλλιευθούν έχει μειωθεί, αλλά γιατί υπήρξε υπεραλίευση και του ε, και του, της υπόγλωσσας και του γάδου και επομένως με τον τρόπο αυτό εξισορροπείται η το αλίευμα και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι θα έχουμε και αηφόρο αλία και εν πάση περιπτώσει θα λαμβάνουμε υπόψη μας και τις συμβουλές των ειδικών. Ο έλεγχος της αλίας λέτε δεν είναι δανέζικος. Όχι, όχι, είναι, είναι όμως βλέπουμε ότι ε, ε, περνούν κάποια ελεύματα από την Δανία στη Γρυλανδία γιατί υπάρχει ειδική συμφωνία άμεσων πωλήσεων ε, από την Γρυλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πρέπει κανείς να διαβάζει προσεκτικά τα πράγματα. Ε, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθειά μας και την εργασία μας έτσι ώστε να απαντηθούν και αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρίστανσεν. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, για τις 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών. Επόμενο σημείο. Δημιουργία κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας. Εμείς τώρα θα παρουσιάσουμε την ε, πρόταση εξ ονόματος της ε, Επιτροπής. Η κυρία Λαϊνέτη, ποιος θα πάρει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πρόταση αυτή στοχεύει ε, στην ε, ευθυγράμμιση της ε, εν λόγω συμφωνίας με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει εδώ τροποποίηση της συμφωνίας για την εξάλληψη παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας. Προβλέπεται εκεί ότι το 2013 θα γίνει μια παρουσίαση στην στο Συμβούλιο και, στην, και στο Κοινοβούλιο σχετικά με, την, τον απολογισμό της συνθήκης Αιγιογιού παράνομης Λευθέρα και Άνοιξης Αλίας. Ε, τον Οκτώβριο ε, θα υπάρξει η έκθεση όσον αφορά την ευθυγράμμιση ε, με, το, με τον κανονισμό ελέγχου και θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Καραμάνη για να σας πει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η κυρία Λενέν προηγουμένως, η πρότασή μας στοχεύει απλώς στην ευθυγράμμιση του κανονισμού για την εξάλληψη παράνομου λαθρέα και άνοιξη με τον κανονισμό λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, βάσει της συνθήκης υπάρχει η πρόβλεψη για μια νέα αντιμετώπιση που χωρίζεται σε κατεξουσιοδότηση και σε εκτελεστικές πράξεις. Το άρθρο 219 παράγραφος 1 για τις κατεξα εξουσιοδότηση και 220 όσον αφορά τις εκτελεστικές εξουσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, άμα τη, εφαρμογή, τη θέση σε ισχύ, ε, ε, εκλήθη να ευθυγραμμίσει τις ε, προηγούμενες αποφάσεις, ε, οι οποίες τώρα βρίσκονται σε διαδικασία συναπόφασης. Οι αλλαγές μας ε, αφορούν μονάχα τις εξουσίες, τι οι οποίες αφορούν και περιέχονται ήδη στον κανονισμό ΙΟΙΟΥ. Μετά από ενδελεχή έλεγχο έχουμε 7 ε, καταλήξαμε σε 7 και 14 αντίστοιχα κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές ε, πράξεις που δεν αλλάζουν όμως την ουσία των αρμοδιοτήτων και ούτως ή άλλως αυτές οι αρμοδιότητες ε, προβλέπονται ήδη στον κανονισμό IUU. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις προτάσεις αυτές. Η πρώτη σχετίζεται με, τον, ε, με το καθεστώς των τρίτων χωρών με τον οποίο δεν υπάρχει συνεργασία. Μετά από πρόταση Επιτροπής, ε, μάλλον ζητήθη απόφαση από το Συμβούλιο, αλλά η απόφαση του Συμβουλίου μετά από αίτημα της Επιτροπής ε, δεν ευθυγραμμίζεται με τα προβλεπόμενα στη δίκη της Λισαβόνας και επομένως η Κομισιόν προτείνει να ε, γίνει εκτελεστική εξουσία αυτή για την ε, Κομισιόν και μια και η φύση αυτής της ε, πράξης αφορά εκτελεστικές αρμοδιότητες να παραμείνει τέτοια και για να απαντηθεί καλά το ζήτημα αυτό θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να παραμείνει η εκτελεστική εξουσία στην Κομισιόν. Δεύτερο σημείο. τα κατεπήγοντα μέτρα προβλέπονται ακριβώς ε, με τον ίδιο τρόπο στον κανονισμό EU λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας θεωρούμε νομίζουμε ότι καλύτερα είναι να μιλήσουμε για temporary measures, για πρόσκαιρα μέτρα. Αλλά ούτως ή άλλως η αλλαγή αυτή δεν αφορά την ουσία. Αποτελεί ευθυγράμμιση όσον αφορά ε, την φύση των μέτρων που έχουν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Ένα τελευταίο σημείο, άρθρο 52. Το άρθρο 52 ε, δίνει ένα γενικό εκτελεστικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Όμως ε, το άρθρο 52 χρησιμοποιήθηκε ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρήση του καθεστώτος για το ε, ειδικό αλευτικό καθεστώς ε, για την αποθήκευση ελευτικών προϊόντων ε, για τα μικρά αλευτικά σκάφη. Επομένως, εδώ προστίθενται τα, η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων από σκάφη τρίτων χωρών. Για να συνεχίσει η λειτουργία αυτής της επιχείρησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υπάρξει ε, κατεξουσιοδότηση πράξη για το απλουστευμένο πιστοποιητικό ΚΑΤΣ ε, και υπενθυμίζω ότι υπήρχε μια ειδική πρόνοια για τα μικρά ε, βιοτεχνικά σκάφη και δεύτερη εξουσία για την προσαρμογή του προγράμματος e Certification σχετικά με το ηλεκτρονικό, προσαρμογή δηλαδή με το ηλεκτρονικό σύστημα τρίτων χωρών. Εδώ ε, προτείνεται ε, συγγνώμη, εκτελεστική, εκτελεστική εξουσία. διότι έχουν ήδη προσαρμοστεί άλλωστε και τρεις εφαρμοστικοί κανονισμοί. 21 Ιουνίου ε, έγινε η έγκριση και αυτομάτως ε, μεταφέρθηκε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή ουσίας, ε, έχουν γίνει μονάχα κάποιες τεχνικές άλλαγες και όπως είπε και η κυρία Λενέ, η ουσία θα ακολουθήσει την, ε, την έκθεση αξιολόγησης που θα σας ε, υποβληθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεβίν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ενημερώσω την Επιτροπή ότι ο συνάδελφος Ρομέρο θα είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα και ελπίζουμε ότι όλοι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην κατάρτιση. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, η κυρία Φράγκα. Κοιτάω και έχω μία αμφιβολία σχετικά με τα έκτακτα μέτρα ε, και τα ειδικά μέτρα, μάλλον τα μέτρα τα εφαρμοστικά σε τρία σημεία. Και θα δούμε πώς αν τα ξαναεξετάσουμε θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε αλλά μπορώ να σας πω σήμερα ότι υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες δεν συμφωνώ απολύτως με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαι διαθέσιμη να το ξανακοιτάξουμε και το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα στα διάφορα. Δεν έχω τίποτα να σας πω. Κυρία Φράγκα, θέλετε κάτι? Θα ήθελα να σας πω ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειλικρινά, η Επιτροπή δεν μας σέβεται καθόλου. Ε, εδώ και πολύ καιρό δεν ε, σέβεται το Κοινοβούλιο και ούτε τη ε, συμφωνία πλαίσιο η οποία προβλέπει ότι οι εκθέσεις και τα βασικά έγγραφα για την εργασία των βουλευτών δεν μπορούν να θεωρηθούν διαβαθμισμένα. Ζητώ δηλαδή μία έκθεση την οποία έχω ζητήσει επανειλημμένος για την τελευταία αντιπροσωπεία σχετικά με τον κανονισμό 1005 ε, για την Νέα που είναι κάποια αντιπροσωπεία ε, η οποία μετέβη το 2011. Επανειλημμένως έχω ζητήσει αυτή την έκθεση και μετά από μία ατέρμονα ανταλλαγή ε, ε, ε, επιστολών με τον πρόεδρο βρίσκουμε ένα έγγραφο το οποίο έχει υποστεί λογοκρισία έχουν ε, διαγραφεί ορισμένα θέματα έχουν διαγραφεί αναφορές σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι εδώ ξεπερνάει τα όρια η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ, αλλά θα χρειαστεί να λάβουμε μέτρα εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθότι εγώ δεν μπορώ να εργαστώ υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν ε, και δεν είναι δυνατόν να μη μου δίδονται έγγραφα που θεωρώ βασικά χωρίς να μου δίδεται καμία εξήγηση. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακόμη πιο περιοριστική σε άλλους τομείς και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε να μπλοκάρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι ότου να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε διότι εγώ δεν μπορώ πλέον να συνεργάζομαι υπό αυτά τα συνθήκας. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Ακούστε με. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητήσαμε συγκεκριμένα σήμερα το πρωί με τους ε, συντονιστές. Ε, κυρία Φράγκα, έχετε απόλυτο δίκιο οι συντονιστές συμφωνούν μαζί σας η κατάσταση αυτή ε, της ελήψεως θεσμικού σεβασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απαράδεκτη. Ε, δεν ε, υπάρχει κανένας σεβασμός και ε, το συζητήσαμε με τους συντονιστές. Πέραν από την ανταλλαγή επιστολών και παράπονα μας λέγεται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα τα μέλη του γραφείου της Επιτρόπου και να σας πω ότι έχουμε προβλέψει μία συνάντηση με την Επίτροπο και κλεισμένων των θυρών. Μία λοιπόν ε, συνάντηση που δεν θα ξεκινήσει με μια μακριά παρουσίαση της Επιτρόπου αλλά εξέταση των θεμάτων που απασχολούν την Επιτροπή μας σε σχέση με την Εκτελεστική Επιτροπή υπάρχουν ορισμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και εμείς θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει την κατάλληλη στιγμή για τη συνάντηση αυτή θα μιλήσουμε για την έλλειψη δεδομένων, την ε, έλλειψη στοιχείων και εγγράφων και θα θέλουμε να λάβουμε μία απάντηση για το τι ε, κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Θα τα ε, διαβάσετε ή στο σημείωμα των συντονιστών και ελπίζω ταχύτερα να καθοριστεί το ραντεβού με την Επίτροπο και αν δεν μας προσφερθεί τίποτα θα ληφθούν αυστηρά μέτρα και ενδεχομένως ένα μπλοκάρισμα όπως το έχει προτείνει ο κύριος Ντέιβις και άλλοι. Ε, το συζητήσαμε όπως σας είπα με τους συντονιστές και ορισμένοι είπαν ότι πρέπει να προσέξουμε για το μπλοκάρισμα που μπορεί ενδεχομένως να είναι αντιπαραγωγικό. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι συντονιστές συμφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δράσουμε ε, θα ζητήσουμε αυτή την συνάντηση με την Επίτροπο και μετά θα δούμε. Συμφωνείτε με αυτό το συμπέρασμα. Ε, αυτή είναι η πρόταση των συντονιστών και τα υπόλοιπα βρίσκονται στο σημείωμα και αν μπορείτε να το δεχθείτε τότε έτσι θα προχωρήσουμε. κυρία Φράγκα. Εντάξει. Οκ. Okay. Έχω όμως και ένα δεύτερο αίτημα που θέλω να υποβάλω θα ήθελα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να προσκληθεί να μας παρουσιάσει τις απόψεις της για τα θέματα λίας, γιατί αυτή η Γενική Διεύθυνση μπορεί να επέμβει στο θέμα του Βιετνάμ για να διαπραγματευτεί μία, για μία συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και θα μιλάμε συνεχώς για τόνο και για ποσοστώσεις και ενδέχεται ε, όλα αυτά να παρεκκλίνουν προς τα θέματα των ναρκωτικών. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν ε, οι σχέσεις με την Ιαπωνία. Είναι δηλαδή ε, θέσεις που έχουν θέματα αλληλείας, περιέχουν θέματα που απασχολούν με την βιομηχανία μας ε, ε, επεξεργασίας της αλληλείας και ε, από τη μία χώρα περνάμε σε άλλες στην Παπουασία, στην Παπούα στη Νέα Γουινέα υπάρχουν θέματα στα οποία προχωρούμε και θα ήθελα η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να έρθει εδώ και να μας πει πόσο θα εξετάσει τα θέματα που αφορούν την αλληλεία ε, και πώς θα τα υπερασπιστεί στις συμφωνίες αυτές ελευθέρου εμπορίου. Ε, δεν νομίζω ότι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου γνωρίζει τα θέματα, η Γενική Διεύθυνση γνωρίζει τα θέματα της Αλίας, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε και να έρθει τουλάχιστον ένας Γενικός Διευθυντής ή ένας Διευθυντής, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη στρατηγική της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου για τις συμφωνίες αυτές. Ευχαριστώ την κυρία Φράγκα. Άλλες παρεμβάσεις. Όντως, το συζητήσαμε χθε. Συμφωνώ. Εχθές είχα την ευκαιρία να συζητήσουμε με την γραμματεία της Επιτροπής και με την Επιτροπή Ίντα και ε, πρέπει να ε, συζητήσουμε ενδεχομένως με τον Γενικό Διευθυντή που ξέρει τι γίνεται και θα ξέρει ίσως περισσότερα και από τον Επίτροπο. Θα γίνει αυτή η προσπάθεια και θα απευθυνθούμε στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου επ' αυτού. Αν δεν έχετε άλλες ε, παρατηρήσεις έχουμε παρουσιάσει κατά κάποιον τρόπο και τις αποφάσεις των συντονιστών. Δεν έχουμε άλλα περίπλοκα θέματα και η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει 19 Σεπτεμβρίου πρωί και απόγευμα στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση.